So, colleagues, we'd to continue our meeting. Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση. Ε, μόλις τοποθετήθηκα ενώπιον των ε, μέσων ενημέρωσης της Ελβετίας, γιατί είχαμε μόλις συζητήσει ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορούσε τη χώρα αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχά του συναδέλφου από την Επιτροπή Ανάπτυξη, ιδίω τον πρόεδρο αυτή, τον κύριο Τομπέ, τον οποίο καλωσορίζω, καθώ και όλου του συναδέλφου τη Επιτροπή ΝΤΕΒΕ. Και θα ήθελα να ε, ε, καλωσορίσω τον κύριο Γκούναρ Βίγκαντ, εκτελεστικό διευθυντή για την Ασία του Ειρηνικού, της ε, ΙΕΔ, που σχεδόν εβδομαδιαίω τον έχουμε πλέον εδώ στη συνεδρία Επιτροπής Εξωτερικών ε, Υποθέσεων. Θα ήθελα επίσης να, να καλωσορίσω τον κύριο Πιέρ Αμιλάτ, Διευθυντή για την Ασία και τη Μέση Ανατολή από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΝΤΕΦΚΟ, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις ε, στο Αφγανιστάν και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χώρα αυτή. Θα ήθελα να ζητήσω από τους ε, προσκεκλημένους μας να μας ενημερώσουν σχετικά με την εφαρμογή στρατηγικής για το Αφγανιστάν, το Αφγανιστάν την ασφάλεια, οικονομικές σχέσεις και την αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα αυτή. Επίσης, ε, θα ήθελα ε, να μας πούν όσον αφορά, το που βρισκόμαστε όσον αφορά την κύρωση από πλευράς κρατών μελών ε, της Συμφωνίας ε, Ανάπτυξης και Συνεργασίας που έχει συναυθεί με αυτή τη χώρα. Ξέρετε ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει εγκρίνει την συμφωνία αυτή φέτος τον Μάρτιο. Αρχικώς είχαμε επίσης προσκαλέσει τον Ρόλαντ Κόμπιε που είναι ο ειδικό απελσταλμένος της Ένωσης για το Αφγανιστάν. Δυστυχώς όμως δεν βρίσκεται εδώ ε, αυτή την εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι οι δύο προσκεκλημένοι μας είναι πλήρως ενημερωμένοι για να μας ε, ενημερώσουν σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Και θα επισέλθουν και στις αρμοδιότητες, στους τομείς αρμοδιότητας του κ. Κόμπιερ. Τελική ε, παρατήρηση από μένα είναι να δώσω καταρχάς το λόγο δηλαδή στον κύριο Τομπέ και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε με την ενημέρωση. Ευχαριστώ, David. Σας ε, χαιρετίζω και για άλλη μια φορά σήμερα, μέλη της ε, ΑΦΕΤ και της ΔΕΒΕ. Είναι πολύ σημαντική χώρα εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν όσον αφορά την ασφάλειά μας και βεβαίως από άποψη πολιτικών σχέσεων που έχουμε αναπτύξει με τη χώρα αυτή ε, βεβαίως υπάρχουν και ε, αναπτυξιακά και ανθρωπιστικά ζητήματα που μας ε, απασχολούν αυτή τη χώρα. Ξέρετε ότι η χώρα αυτή είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραλήπτες ε, βοήθειας ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής. Η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2002 έχει παράσχει πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα σε μορφή ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας και ε, έχουμε πλέον τη συμφωνία με, την, ε, με, την, ε, Αυγαν, με το Αφγανιστάν όσον αφορά και στο πλαίσιο της κοινή γεωργικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πλέον τονίζεται ότι ε, στόχος είναι η ενίσχυση της γεωργίας του Αφγανιστάν, η ε, επίτευξη της αυτάρχειας της χώρας. Θέλουμε λοιπόν από τους προσκεκλημένους μας να μάθουμε πώς προχωρούν τα πράγματα ε, υπό το φως και της περίπλοκης κατάστασης της πολιτικής και από άποψη ασφάλειας. Η κατάσταση αυτή έχει ε, δυσκολέψει λόγω του, ε, της απότομης αύξησης του επίπεδου φτώχειας, ε, του ποσοστού φτώχειας από 38% σε 2015 σε 55% το 2017 ε, είναι μια δύσκολη εικόνα αυτή και από την άποψη της αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχεται. Αυτά θέλουμε να συζητήσουμε. Πρόεδρος της ΑΦΕΤ, ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκούναρ Βίγκαντ για 7 έως 10 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι, τους κυρίους Προέδρους ζητήσατε για πληροφορίες σχετικά με τη Συμφωνία Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης ε, η οποία βρίσκεται υπό καθεστώ προσωρινή εφαρμογή από το Δεκέμβριο του 2017. 17 κράτη-μέλη έχουν κυρώσει τη συμφωνία αυτή. έω ότου ε, κυρωθεί και από του 27 και ή 28 δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε πλήρη εφαρμογή αυτής της ε, συμφωνίας. Ωστόσο, μας έχει βοηθήσει να διαρθρώσουμε και να δομήσουμε την συνεργασία μας με το Αφγανιστάν. Αυτή τη βδομάδα ε, ε, μόλις ολοκληρώσαμε ε, μια μακρά, ε, μια μεγάλη συνάντηση των Γενικών Διευθυντών από τις πρωτεύουσε και έγινε και μια συνεδρίαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας στη σύνοδο που έγινε την Δευτέρα. Πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή λοιπόν για τη σταθερότητα της περιοχής καθώς και για τις μελλοντικέ εξελίξεις ε, και τις σχετικές δυνατότητες, ε, τις δυνατότητες ανάπτυξης του Αφγανιστάν. Μένεται ο εμφύλιος πόλεμος, αναζωπηρώθηκε κιόλας και δημιουργούνται νέες προκλήσεις για τη μετάβαση στην ειρήνη συνολικά για τους πολίτες της χώρας. Πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε ότι θα αξιοποιηθεί η νέα ορμή ε, υπέρ μια ειρηνευτική διαδικασία και να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την διεθνή διαδικασία, την διεθνή ειρηνευτική διαδικασία. Ε, και όχι μόνο να ε, αποτελεί έναν πάροχο αναπτυξιακής βοήθειας βεβαίως αυτή η αναπτυξιακή βοήθεια είναι πολύ σημαντική, δεδομένων και των ποσοστών που αναφέρατε εσεί όσον αφορά την φτώχεια. Η χώρα ε, κατά 55% εξαρτά τις ε, δαπάνες του προϋπολογισμού από ε, ε χορηγίες ε, και στήριξη χρηματοδοτική από το εξωτερικό. Πολλά, λοιπόν, πολλές λοιπόν προσδοκίες υπάρχουν στο πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις δημοκρατικές δυνάμεις του Αφγανιστάν. Το ίδιο και από τη δική μας πλευρά βεβαίως. Έχουμε πολλές προσδοκίες. Τα τελευταία χρόνια έχουμε διαδραματίσει θετικό ρόλο. Υπερασπιστήκαμε παρά τις απειλές για την ασφάλεια, παρά τις ε, προσπάθειες ειρήνευσης με τους Ταλιμπάν από τις ΗΠΑ μέσω διμερών ε, επαφών ότι πρέπει να διεξαχθούν εκλογές και να τηρηθεί το Σύνταγμα, ακόμα και όταν πολλοί ε, εμπλεκόμενοι φορείς και ενδιαφερόμενοι είχαν εγκαταλείψει κάθε τέτοια ιδέα. Το Σεπτέμβριο του 2019 οι εκλογές που διεξήχθησαν ήταν τεράστιο επίτευγμα και απέδειξαν τον υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας της ε, αφγανικής δημοκρατίας. Από τεχνικής και άποψης και άποψης, από άποψης ασφάλειας ήταν οι καλύτερα διοργανωμένες εκλογές που έχουν διεξαχθεί ποτέ στη χώρα, αν και το ποσοστό συμμετοχής ήταν απογοητευτικό. Μόλις το 20% των ψηφοφόρων προσήλθε στις κάλπες και αυτό Επίση, ε, επίσης ε, ένα στοιχείο των εκλογών αυτών ήταν ότι χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά ε, οι συσκευές βιομετρικής ταυτοποίησης των ψηφοφόρων. Οι διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνηση ε, αναμένονται να γίνουν στο τέλος του τρέχοντος μηνός αν και αναβάλλεται αρκετά αυτή η ημερομηνία. Ελπίζουμε η καταμέτρηση των ψήφων να ολοκληρωθεί ε, σύντομα γιατί ήταν και, ε, χρησιμοποιήθηκε και ένα σύστημα ευρωπαϊκό ε, όσον αφορά τις ε, συσκευές ταυτοποίησης με βιομετρικά στοιχεία για να αρθούν προβλήματα που είχαν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν σχετικά με νοθεία. Ο πρόεδρος, ε, ωστόσο, χρειάζεται το 50% των ψήφων στον πρώτο γύρο. Κάτι τέτοιο δεν επετέφθη. άρα θα γίνει δεύτερος γύρος ε, του επόμενου μήνε. Από τον δεύτερο γύρο και έπειτα ελπίζουμε πια να ε, οδηγηθούμε σε πολιτική σταθερότητα και να ε, πρέπει να συμβάλλουμε κι εμείς ε, στο να προχωρήσουμε σε μια έφτακτη διαδικασία, στο να υπάρχει ένα νόμιμος πρόεδρος και μια νόμιμη κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να προσέλθει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν, οι οποίε μπορούν να ξεκινήσουν αφότου καταλήξουν οι Ταλιμπάν με τους ΗΠΑ σε συμφωνία. Η κυρία Μογκερίνη φέτο ε, ε, στι αρχέ του χρόνου είχε πάει στο Αφγανιστάν και ο στόχος ήταν και εκλογές και ειρήνευση. Και οι δύο στόχοι πρέπει να επιδιωχθούν. Στην Υπουργική Διάσκεψη της Γενέφης του, το Δεκέμβριο του 2018 η κυρία Μογκερίνη είχε ε, ε, δώσει και κάποια κίνητρα για την υπέρβαση χρόνιων προβλημάτων του Αφγανιστάν όσον αφορά την ένταξη, την ένταξη πρώην μαχητών, ε, ε, την ειρήνευση, την ε, κοινωνική ευημερία. Πέντε συγκεκριμένα σημεία είχε παρουσιάσει και εμείς εξειδικεύσαμε τα πέντε αυτά σημεία σε μια συγκεκριμένη προσέγγιση για να ισχυροποιήσουμε και όχι να διαβρώσουμε βεβαίως την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία 18 χρόνια και να εξασφαλίσουμε τη συνταγματική συνέχεια. Υπάρχουν λοιπόν θέσεις αρχής τις οποίες υπηρετούμε συστηματικά και με συνέπεια, κάτι που δεν μπορούμε να πούμε για όλους τους εμπλεκόμενους ε, φορείς ε, στο διεθνές στερέωμα. Με τους εταίρους μας λοιπόν ε, συνεχίζουμε να δραστηριοποιούμαστε όχι μόνο για, ε, για την υποστήριξη, όχι μόνο, ε, για την υποστήριξη των πολιτών, αλλά όχι μόνο από ευρωπαϊκής πλευράς, ώστε να πάρει έναν χαρακτήρα πιο διεθνή και παγκόσμιο η στήριξη αυτή. Οι άμεσες ε, συνομιλίες μεταξύ Ταλιμπάν και ΙΠΑ αποτελούν πολύ κρίσιμο στοιχείο, βραχυπρόθεσμα, γιατί θα οριστικοποιήσουν τους ε, όρους της συμφωνίας αποχώρησης των Αμερικανικών στρατευμάτων καθώς και τις δεσμεύσεις που θα αναλάβουν οι Ταλιμπάν. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι κάθε τέτοια συμφωνία θα πρέπει να συνοδεύεται από ε, μείωση των ε, ε βιοπραγιών και ε, να οδηγεί σε ανακοχή και τελικά σε πλήρη εκεχηρία. Το σημαντικότερο λοιπόν ε, βραχυπρόθεσμο συνοδευτικό μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση είναι ότι θα πρέπει άμεσα να σταματήσει το φαινόμενο να υπάρχουν άμαχοι νεκροί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει την σημασία ε, την, ε, που έχει να συμπεριλαμβάνει η διαδικασία αυτή της ειρήνευσης όχι μόνο την κυβέρνηση αλλά και την κοινωνία των πολιτών, τον ίδιο τον αφγανικό λαό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η κυβέρνηση του Αφγανιστάν είναι σημαντικός εταίρος όσον αφορά την ε, προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημιουργικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των γυναικών που τόσοι αγώνες έχουν γίνει για να κατακτηθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από την πρόσφατη ε, απόσυρση του ε, Trump. Τραμπ ε, και, το, και τις σχετικές ανακοινώσεις του στο Twitter ανέλαβε τις υποχρεώσεις ε, ε, της και στη Μόσχα σε συνάντηση που έγινε ανάμεσα στο Αφγανιστάν, της είπα και τη Ρωσία στην οποία συμμετείχαμε και εμείς ε, σημειώσαμε πρόεδρο, αντίστοιχη, ε, πρόοδο, αντίστοιχη ε, συνάντηση θα γίνει το επόμενο διάστημα και στο Πεκίνο υπό την αιγίδα της Κίνας. Αυτή δεν είναι η ίδια η διαπραγματευτική διαδικασία, αλλά όλες αυτές οι εκδηλώσεις μπορούν να βελτιώσουν το κλίμα μεταξύ των δύο αφγανικών πλευρών, ώστε να ξεκινήσουν πραγματικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό στο Όσλο και αν μου δώσετε τη δυνατότητα στο, ε, λίγο αργότερα μπορώ να επισέλθω και σε λεπτομέρειες σχετικά με τα όσα αφορούν τους περιφερειακούς μας εταίρους, αλλά προς το παρόν σταματώ ε, για να δώσω το λόγο στον συνάδελφο από την ε, Γενική Διεύθυνση Ντεύκο. Yes, uh, two really. The first one on the state of play. Δύο σημεία. Πρώτον, κατάσταση πραγμάτων ε, συνεργασία με το Αφγανιστάν και δεύτερον στραμμένη προς το μέλλον ε, ποιες είναι οι προσπάθειες ε, για, για τα στοιχεία τα οποία ονομάζονται rules of engagement. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ ε, ο όρος αυτός, αλλά πάντως αφορά τις ε, διαδικασίες της ειρήνευσης. Όσον αφορά την κατάσταση των πραγμάτων, το Αφγανιστάν ε, είναι το πιο ευρύ, ο πιο ευρύς φάκελος συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο και βεβαίως ε, ε, εμείς πάντα προσπαθούσαμε για την ειρήνευση και την οικοδόμηση ε, του κράτους, λαμβάνοντας υπόψη το, περιεχο... το, το περιφερειακό κόντεξτ Αυτή τη στιγμή ε, και στο παρόν πι ε, έχουμε αφιερώσει περίπου 1,4 εκατομμύρια, δηλαδή 200 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος ε, τομείς ε, προτεραιότητες ε, είναι η δημοκρατία, η σταθερότητα και η ειρήνη. Δεύτερον, βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση. Και τρίτο είναι η προμήθεια βασικών υπηρεσιών στους και παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και βεβαίως έχουν ξεκινήσει διάφορες δράσεις συντονισμένες το 2010 για ε, να σας δώσω μια ιδέα για τα προγράμματα τα οποία ξεκίνησαν ή θα ξεκινήσουν. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την πρόθεση του εμπορίου στο Αφγανιστάν, δηλαδή καλύτερη ε, σύνδεση της χώρας με τους ε, με τους γείτονες. Το δεύτερο είναι η, η υποστήριξη των ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων, agribusiness γενικά, 30 εκατομμύρια δίνουμε σε αυτό το ετήσιο πρόγραμμα. Πρόκειται για μια ανάγκη η οποία ταυτοποιήθηκε πριν από πολλά χρόνια ήδη και από την Παγκόσμια Τράπεζα. Ε, επίσης, ε, η προώθηση και η υποστήριξη των λεγόμενων Citizens Charter που αφορά βασικές υπηρεσίες που ε, μπορούν και πρέπει να παρέχονται ε, στην κοινότητα. Εδώ δίνονται 17 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως, η ειρήνη, ε, δημιουργία θέσεων εργασίας και αύξηση του εισοδήματος, αυτά είναι οι μεγάλες προτεραιότητες. Διανύουμε μια περίοδο αβεβαιότητας ε, όσον αφορά τη διαδικασία ειρήνευσης, αλλά ε, είναι ευρία η συνένεση όσον αφορά τις βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθήσουμε προετοιμαζόμενοι για το μέλλον. Ε, δηλαδή ε, είναι σαφές ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα πισωγύρισμα όσον αφορά τα όσα έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα και όσον αφορά και τις μεταρρυθμίσεις, προστασία των παιδιών, ισότητα φύλων, όλα αυτά και όλες οι πρόοδοι που έχουν γίνει ε, στα θέματα αυτά ε, στο Αφγανιστάν δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να ε, πάνε πίσω, να υποχωρήσουν λόγω του ότι δεν έχει προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία. Όπως είπε και ο συνάδελφος μου προηγουμένως, είναι σαφές ότι το Αφγανιστάν και τώρα, αλλά και για πολύ καιρό ακόμα, θα, ε, εξαρτάται από την εξωτερική ε, βοήθεια. Πέρα από οποιασδήποτε καλές προσπάθειες έχει καταβάλει ο Υπουργός Οικονομικών ε, του Αφγανιστάν, η θέση του Δουνουτού, καθώς επίσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ε, είναι απόλυτα σαφής και πολύ αυστηρή ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε εξωτερικό δανεισμό η χώρα. Και εμείς οι ίδιοι έχουμε δώσει ε, βοήθεια στη χώρα από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως άλλωστε κάνουν και οι περισσότεροι δωρητές, που ε, προχωράνε είτε σε άμεσες δημοσιονομικές ε, βοήθειες, είτε μέσω του RDF, δηλαδή το καταπίστευμα του Αφγανιστάν για την επανίδρυση. όλη η αρρωγή που παρέχεται στην ε, χώρα από τους συναδέλφους ε, της ε, ΕΚΟ, δηλαδή η ανθρωπιστική βοήθεια δεν πρέπει να υποτιμάται με κανένα τρόπο. Πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ ισχυρή η περιφερειακή διάσταση των όσων κάνουμε στο Αφγανιστάν ε, αυτή η περιφερειακή διάσταση προωθήθηκε, υπογραμμίστηκε στη διάρκεια της διάσκεψης των δωρητών ε, που οργανώθηκε στην, ε, στις Βρυξέλλες ήδη από το 2016 κυρίως όσον αφορά και τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Μισό δις ε, ευρώ έχει ήδη επενδυθεί ε, όσον αφορά την ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων, ε, το διασυνοριακό εμπόριο και την επένδυση, ενέργεια και περιβάλλον, ε, μεταφορά και συνδεσιμότητα ψηφιακή και τέλος πολιτισμός και εκπαίδευση και με το γειτονικό Πακιστάν ιδιαίτερε σχέσεις έχουν αναπτυχθεί όσον αφορά το τελευταίο αυτό θέμα. Αυτό που θέλουμε είναι να γίνουν περισσότερες επενδύσεις έτσι ώστε το Αφγανιστάν να πάρει μια ισχυρή θέση ε, στο περιφερειακό του περιβάλλον. Να πω και δύο λόγια ε, για, την, ε, για τις συμβάσεις που έχουν γίνει όσον αφορά την βελτίωση της κατάστασης στη χώρα. Έχουμε καλές state building contracts ε, είχαμε ένα πρώτο από το 16 μέχρι το 19 και ένα νέο μετά από τη διάσκεψη της ε, ε, Γενέβης, διάσκεψη των δωρητών, που θα καλύψει τα τρία επόμενα χρόνια. Επομένως έχουμε πέντε έτη συγκεκριμένων και προβλέψιμων χορηγιών προς το Αφγανιστάν έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές δημοσιονομικό εργαλείο ε, έτσι ώστε να πληρώνονται τα πάγια κόστη, να πληρώνεται η εκπαίδευση, να, να χρηματοδοτούνται οι απαραίτητες πολιτικές συμπεριλαμβανομένες και της κοινωνικής ε, πολιτικής. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι λοιπόν με αυτό. και οπωσδήποτε έχει υποστηρίξει την ε, εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη αυτή η διαδικασία. Ε, όσον αφορά την μετανάστευση και τις υποχρε... τους υποχρεωτικούς ε, εκτοπισμούς ε, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο πάντοτε μας απασχόλησε, είναι δυναμικό, είναι εξελισσόμενο, αφορά και τους γείτονες, ξέρετε ειδικά με το Πακιστάν είχαμε πολλές επιστροφές από την Τουρκία, περίπου 200 επιστροφές ανά ημέρα που αφορούν την Καμπούλα αλλά και άλλες ε, ε, πόλεις. Και εμείς υποστηρίζουμε αυτήν την διάσταση της μετανάστευσης, ενώ ταυτόχρονα ε, προσπαθούμε να ξαναεντάξουμε τους ανθρώπους αυτούς στον οικονομικό ιστό της χώρας. Ε, βεβαίως εμείς εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε το Αφγανιστάν παράλληλα με την ειρηνευτική διαδικασία, ε, προσπαθώντας ανα πάσα στιγμή να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε, κυρίως ε, κυρίως όσον αφορά την άμεση παροχή ε, ανθρωπιστικής βοήθειας ε, και όσον αφορά και την παροχή υπηρεσιών ε, σε πιο απομακρυσμένες περιφέρειες βάσει και αυτού του People Charter που ανέφερα προηγουμένως και που έχει δώσει αρκετά αποτελέσματα μέχρι τώρα. Τούτων λεχθέντων βεβαίως ε, προσπαθούμε να ε, μελετήσουμε καλύτερα και τις λεγόμενες rules of engagement, κανόνες εμπλοκής. κατά την άποψή μας ε, θα πρέπει να ληφθούν ε, ε, σωστά υπόψη απέναντι στο Αφγανιστάν και χωρίς όμως να αποτελούν προϋπόθεση. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει πρώτα συμφωνία μεταξύ των Αφγανών. Έχουμε όμως και κάποιες ενδείξεις για σοβαρά στοιχεία για μας. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, δηλαδή καμία οπισθοχώρηση, οπισθοδρόμηση σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις και σε σχέση με ό,τι έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα ε, υποστήριξη δημοσιονομική, μακροοικονομικές πολιτικές που δεν μπορούν όμως να ολοκληρωθούν χωρίς διαφάνεια του προϋπολογισμού και χωρίς την εφαρμογή ορθών ε, πολιτικών καθώς επίσης και ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι γνωστά ε, στην όποια μελλοντική κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Επίσης είναι σαφές ότι έχει ουδέτερη στάση η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζει τη χώρα, δεν υποστηρίζει τη μία ή την άλλη κυβέρνηση. Δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί το ενδιαφέρον έγκυται στην ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τους δύο κυρίους για τα εισαγωγικά τους ε, σχόλια, παρατηρήσεις. Ε, μπορούμε να συζητήσουμε τώρα τις ε, παρουσιάσεις αυτές. Άννα Πρώτα απ' όλα που στην προηγούμενη θητεία βεβαίω υπήρξε εισηγήτρια επί του Αφγανιστάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους ε, Γενικούς Διευθυντές για την ενημέρωσή τους, για την εισήγησή τους, για την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Ελπίζω να κυλήσει ομαλά η διαδικασία της επικύρωσης ώστε να μπορέσουμε σύντομα να εφαρμόσουμε την πλήρη συμφωνία. Όλοι μας ε, γνωρίζουμε ότι αποφασίζουμε, μάλλον ότι αντιμετωπίζουμε μια αποφασιστική στιγμή. Διερχόμαστε μιας κρίσιμης στιγμής αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε πόσο ευάλωτη είναι η ισορροπία και τα οποιαδήποτε λανθασμένα βήματα θα μπορούσαν να διαταράξουν αυτήν την ευάλωτη ισορροπία. Φυσικά, διερωτώμεθα και για το επίπεδο της αμερικανικής δέσμευσης γιατί εξ όσων γνωρίζω υπάρχουν κάποιες σκέψεις αποχώρησης και υπάρχουν και κάποιες πτυχές εσωτερικού συσχετισμού δυνάμεων. Πώς θα εκτιμούσατε εσείς την δύναμη που έχουν σήμερα οι Ταλιμπάν η, η ενεργητική τους ικανότητα ποια είναι. Πώς αξιολογείται τις πιθανότητες να επιτύχουμε θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε την κυρία Φωτίγκα. Ο κύριος Νάρτ παρακαλώ. Ε, παρακολούθησα με προσοχή πρόεδρε. τι εισηγήσεις σχετικά με δραστηριότητες, θα έλεγα με επιθυμίες γιατί η πραγματικότητα στο έδαφος είναι ότι έχουμε μια χώρα αποτέλεσμα της ιστορίας της όπου οι μόνες ασφαλείς ζώνες είναι συνοριακές με Ουσμπεκιστάν και Τατζικιστάν των οποίων ηγούνται ε, αρχηγοί γενοκτονιών που ξεχνούμε συνήθως τις γενοκτονίες που έχουν διαπράξει στο παρελθόν επίσης κοντά στον Μπαμπιγιάρ που ελέγχονται οι ζώνες από άλλους εξωτερικούς. Κατά τα άλλα μιλούμε για ε, ε, περιοχές ελεγχόμενες από τους Παστού, δηλαδή υπό τους Ταλιμπάν, οι οποίοι έχουν γνωστές ε, ιδεολογικές βαρβαρικές προσεγγίσεις, αλλά αποτελούν την πραγματικότητα. Χωρίς τους Ταλιμπάν ή εναντίον τους λύσεις δεν υπάρχει. Και μιλώντας για την κυβέρνηση του Αφγανιστάν μήπως μιλούμε πέρα από τις επιθυμίες μας δηλαδή απλώς για το Δήμο της Καμπούλ γιατί πέραν της Καμπούλ καμία επιρροή δεν έχει. Όταν είχαμε ισπανικές ε, ε μονάδες κοντά στην Χεράτ όπου έπρεπε να βοηθήσουν στην ε, κατασκευή σχολείων, ε, διόδων άρδευσης δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν καν την συνεργασία των τοπικών φορέων στις ζώνες που αναπτύσσονται οι δικές μας στρατιωτικές δυνάμεις. Ε, έχουμε κατακερματισμένες διαπραγματεύσεις στο Κατάρ μεταξύ των Ταλιμπάν και των ΙΠΑ ε, ε, γιατί οι Ταλιμπάν έναντι της κυβέρνησης της Καμπούλ δεν έχουν την παραμικρή εμπιστοσύνη. Οι μυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν έχουν άμεση και στενή σχέση με τους Ταλιμπάν. Δηλαδή θα έπρεπε να βγούμε από την φαντασιακή πραγματικότητα και να πάμε στην πραγματικότητα. Και η ερώτησή μου είναι απλή. Ποια εναλλακτική έχουμε απέναντι στην τερατώδη αλλά μάλλον απαραίτητη διαπραγμάτευση με τους Ταλιμπάν. Όταν το σημείο της σημεία επιστροφής ακούω να λέτε ότι είναι ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, συμφωνώ δηλαδή μαζί σας, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι σε οποιαδήποτε περιοχή εκτός της Καμπούλ η παράδοση της χώρας ε, δεν είναι ακριβώς αυτή, να σας το πω έτσι. Επομένως δεν μιλούμε για πολιτικές προσδοκίες, μιλούμε για επιστημονική φαντασία εδώ. Σας ευχαριστούμε, Χαβιέρ. Dominic Μπίλντ, Aldi, παρακαλώ. Ευχαριστώ, ε, κύριε Πρόεδρε η στρατιωτική υποστήριξη από τη δεκαετία του 2000 πολεμική επιχείρηση από τις δύο φιλόδοξες ένα δισεκατομμύριο το χρόνο μαστίζει και παραπάνω και όλα αυτά για να είμαστε σήμερα σε τραπέζι διαπραγμάτευση με τους Ταλιμπάν και μπροστά σε ένα κατεστραμμένο αποτυχημένο κράτος πρόκειται για μια κατάσταση που μας λέει όσα χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε σχετικά με διεθνείς επιχειρήσεις ανατροπής καθεστώτων χωρίς να υπάρχει αναλλακτική λύση, χωρίς να υπάρχει σχεδιασμός, πέρα συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων όπως η δική μας που είχε αντιταχθεί σε αυτές τις ε, διεθνείς επιχειρήσεις. Έχουμε 17.000 Αφγανούς ε, πρόσφυγες μετανάστες προς την Ελλάδα, για παράδειγμα. Το 2016 είχαμε μια ε, συμφωνία που υπεγράφει και η οποία υποτίθεται ότι διευκόλυνε την επιστροφή στις χώρες προέλευσης, αλλά στην πράξη τίποτα τέτοιο δεν συμβαίνει. Έχετε εκτιμήσει ή αξιολογήσει την επιδείνωση της κατάστασης ε, της προσφυγικής, δηλαδή των προσφυγικών ροών από το Αφγανιστάν προς την Ευρώπη και πώς φαντάζεστε ότι μπορούμε να διευκολύνουμε επιστροφή προς τη χώρα αυτή υπό τις συνθήκες της απαράδεκτης που επικρατούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Μπίλντ. Ο κύριος Γκάλα. Ευχαριστώ. Έχω την ε, αίσθηση ότι είχαμε βασιστεί σε διαπραγματεύσεις που αν είχαν ολοκληρωθεί επιτυχώς ε, θα έδιναν μέρος της εξουσίας επί της χώρας και στους Ταλιμπάν. Ότι θα ε, σταματούσαν οι συγκρούσεις, όμως ότι θα είχαν επιρροή οι Ταλιμπάν και στην κυβέρνηση. Αυτό τελικά δεν έγινε και αυτό δημιουργεί κίνδυνο και φόβους ότι θα συνεχιστεί ο πόλεμος σε μεγάλο μέρος της επικράτειας της χώρας. Αν θέλουμε όμως τελικά να οδηγηθούμε σε ειρήνευση, ε, θα πρέπει ε, με κάποιο τρόπο να συμμετάσχει στη διαδικασία αυτή και η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι Αμερικάνοι με τους Ταλιμπάν και εκ μέρου τη δύση οι Αμερικάνοι τους υπόσχονται διάφορα πράγματα όπως για παράδειγμα ότι δεν θα ξαναγίνει χώρα ε, λίκνο της τρομοκρατίας ε, και συμμοριών και τους ανατίθεται ε, στην κυβέρνηση του Αφγανιστάν με συμμετοχή και των Ταλιμπάν ότι θα τα λύσουν μόνα τους αυτά τα πράγματα. Και όλα αυτά ε, καλούμαστε εμείς να τα αποδεχτούμε διότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος ε, όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, στην εκπαίδευση κτλ. Το ερώτημα που τίθεται για μένα είναι σε ποιο βαθμό θα ήμασταν κι εμείς, ε, αν πράγματι τα πράγματα έρθουν έτσι, να συνεχίσουμε να δίνουμε χρηματοδότηση στη χώρα αυτή. Πώς θα μπορούμε να χρηματοδοτούμε μια χώρα ε, στην οποία, στις στην κυβέρνηση θα συμμετέχουν οι Ταλιμπάν. Πώς θα μπορούμε να κάνουμε προγράμματα έργα σε μια τέτοια χώρα γιατί νομίζω ότι γενικότερο στόχο μα, όλα αυτά τα χρόνια ήταν η χειραφέτηση των γυναικών, των παιδιών κτλ. Όλα αυτά δηλαδή ήταν στόχοι οι οποίοι προφανώ δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ε, με συμμετοχή, με κυβέρνηση στην οποία θα συμμετέχουν οι Ταλιμπάν. Πώ θα μπορέσουμε δηλαδή να γυρίσουμε και να πούμε απλά ότι εντάξει καλά μια χαρά δεν πειράζει και οι Ταλιμπάν μέσα. Πώς μπορούμε μια τέτοια προοπτική εμείς να την ε, αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Άλλους δύο μιλητές θα ακούσουμε και συνέχεια θα δώσω λόγο τους, ε, στους δύο προσκεκλημένους μας. Για το ID, ο κύριος Τσίμνιοκ έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ε, ο κύριος Τσίμνιοκ, Herr Τσίμνιοκ. Συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, δεν ήξερα ότι είστε Γερμανός. Δεν πειράζει, όλοι ίσοι είμαστε. Έμαθα από τον τύπο ότι εδώ και τέσσερις εβδομάδες 300 Αυγανοί έχουν διασχίσει τα σύνορα ε, Ιράν προς την Τουρκία και ότι η Τουρκία έχει αντιμετωπίσει σοβαρότατα προβλήματα. Από την άλλη πλευρά ακούω ότι υπάρχει, υπάρχουν επιστροφές από την Τουρκία και προς το Αφγανιστάν. Κάτι που δεν μου ακούγεται και πολύ πιθανό. Διότι αυτή τη στιγμή η, το Ιράν μειώνει τον αριθμό των Αφγανών προσφύγων που φιλοξενεί. Εγώ ε, θα ήθελα να μάθω αυτή η πληροφορία περί 200 πληροφοριών ε, ατόμων που μας ε, δώσατε εσείς είναι αξιόπιστη γιατί αξιόπιστη είναι και η πληροφορία που σας δίνω εγώ για 300 ανθρώπους. Και επίση, το ερώτημα είναι, ποια είναι η κατάσταση ασφαλείας στο Αφγανιστάν. Υπάρχουν ε, περιφέρειες της χώρας στην οποία οι Ταλιμπάν δεν έχουν καθόλου έλεγχο, καμία δύναμη. Μήπως θα μπορούσαν οι επιστροφές να γίνονται σε αυτές τις ε, περιοχές. Αυτό θα ήταν μια ρεαλιστική λύση. Διαφορετικά αυτές οι ροές θα έρθουν στην Ευρώπη και από εκεί και πέρα θα χάσουμε κάθε έλεγχο. Όπως ακούστηκε, τα ποσοστά των επιστροφών είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ε, ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε ε, με αυτόν τον τρόπο να ανακατευθύνουμε τις μεταναστευτικές προσφυγικές αυτές ροές προς αυτές τις περιφέρειες ώστε να μην έρθουν προς την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Λέω πρόεδρος, η κυρία Μπέντελε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να Μα ε, δώσετε ορισμένε προφορές σχετικά με του φορεί που αναλαμβάνουν την αναπτυξιακή βοήθεια, την παροχή αυτή τη αναπτυξιακή βοήθεια. Ποιοι είναι οι βασικότεροι παίκτε σε αυτή τη διαδικασία, ποια είναι η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Και συνολικά ε, πείτε μα ε, κάποια λόγια και για την ανθεκτικότητα τη κοινωνία των πολιτών στο Αφγανιστάν. Σε ποιο βαθμό τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να χειραφετηθεί η κοινωνία των πολιτών και να ανεξαρτητοποιηθεί από διάφορα πιο παραδοσιακά αν θέλετε στοιχεία και σε ποιο βαθμό έχει καταφέρει να αποτελέσει έναν αυτόνομο ε, φορέα. Ο κύριος Σικόρσκι, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, να σας πω ότι ξεκίνησα ήδη το 1996 να πηγαίνω στο Αφγανιστάν ε, όταν ήταν υπό, ε, σοβιετικής, υπό σοβιετική κατοχή. 79, when they came to the assistance of regime that was about to και τότε υπήρχε ένα κομμουνιστικό καθεστώς το οποίο ήταν έτοιμο να ε, καταρρεύσει. Εν πάση περιπτώσει, ε, νομίζω ότι ε, τότε βοηθήσαμε τους Αφγανούς που ούτως ή άλλως ήθελαν την κατάρρευση αυτού του καθεστώτες, αλλά έγιναν τότε πολλά λάθη. Πρώτα απ' όλα δεν καταφέραμε να υποστηρίξουμε τους αντικομουνιστές ε, Αφγανούς να επανοικοδομήσουν το κράτος ε, και ε, όταν, όταν νικήσαμε τους Ταλιμπάν βάλαμε τα δικά μας στρατεύματα μέσα. Το 11 οι Ταλιμπάν ε, στην ουσία ε, μέσα σε έξι εβδομάδες και με μεγάλη ευκολία ιτήθηκαν ε, με κάποια χρήματα και κάποιες αεροπορικές επιδρομές. Εντάξει, όμως τότε ίσως λόγω ελλειπού συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων θεσμών δεν καταφέραμε να δώσουμε πραγματικά λύσεις στα προβλήματα. Σε ορισμένες περιφέρειες δεν έφτανε ποτέ η αναπτυξική βοήθεια. Και γιατί αυτό, γιατί για δικούς μας λόγους δεν καταφέραμε να έχουμε καλή συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μόνη λύση στο Αφγανιστάν ήταν να ζητήσουμε από το ε, ΝΑΤΟ να περιφρουρεί τις PRT, αυτές δηλαδή τις Provisional Reconstruction Teams, ε, και ε, όμως το ΝΑΤΟ δεν μπόρεσε να συνεργαστεί λόγω διαφωνιών μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας λόγω της Κύπρου. Και μετά από 17 χρόνια ε, δεν καταφέραμε τίποτα περισσότερο από ότι η Σοβιετική τότε και οι φιλοευρωπαίοι ε, Αυγανοί τελικά ε, πλήρωσαν και πληρώνουν ένα πολύ υψηλό βαρύ τίμημα. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στους δύο μιλητές μας, παρατηρήσει εκτός μικροφώνου δεν ακούν οι διερμηνείς. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, πρέσβη του Αφγανιστάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Ναζάλ Αλ Αλ-Ασάνι. Κύριε Γκούναρ Βίγκαντ, έχετε το λόγο. Η πρώτη μου αντίδραση σε αυτά τα πολλαπλά σχόλια είναι ότι θα πρέπει πιο συχνά να συζητούμε για το θέμα του Αφγανιστάν. Είναι μια χώρα ε, προς την οποία έχουμε μεγάλη δέσμευση και το ΝΑΤΟ και το, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι εταίροι ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και Πρόκειται για μια χώρα στην οποία δείχνουμε μεγάλο ε, ενδιαφέρον και σίγουρα ε, τα θέματα ασφάλειας και μαζικής μετανάστευσης είναι ε, κάποια απορρέοντα στοιχεία τα οποία ιδιαίτερως μας απασχολούν και τα οποία ανέφεραν ορισμένοι μεταξύ ημών. Είναι γεγονός ότι ο Άισις ε, μπορεί να έχει ιτηθεί σε κάποια, σε κάποια άλλα μέρη, αλλά φαίνεται ότι οι ξένοι μαχητές ε, του Τζιχάντε και μέλη του Άισις φαίνεται να ανασυστήνονται ε, στο Αφγανιστάν. Επομένως πρέπει να παραμείνουμε δεσμευμένοι, αλλά και ακόμα περισσότερο να δεσμευτούμε στο Αφγανιστάν. Έχουμε βεβαίως ε, απέναντί μας και τις ε, θεσμητές προσδοκίες ε, των Αφγανών. Και πρέπει να σας πω ότι όλοι θέλουν να βοηθήσουν το Αφγανιστάν εκτός από την Ιαπωνία, τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία και τα Ηνωμένα Εμμυράτα και Αραβικά Εμμυράτα και η Κίνα κλπ. Ωστόσο νομίζω ότι πλέον οι Αφγανοί έχουν κουραστεί από τον πόλεμο, έχουν κουραστεί από τον εμφύλιο μόιλο, πόλεμο, έχουν κουραστεί από ε, τις, τους εκτοπισμούς ε, και την μετανάστευση. Ναι, είναι γεγονός ότι υπάρχουν επιστροφές ε, από το Πακιστάν, όχι πάντα εθελούσιες, αλλά και από το Ιράν όπου η κατάσταση οικονομική διαρκώς χειροτερεύει και ξέρουμε τους λόγους. Ε, δεκάδες ε, χιλιάδες ε, επιστρέφονται από το Πακιστάν, ενώ οι αριθμοί επιστροφών από, την, από το Αφγανιστάν είναι πολύ μικρότεροι. Είναι γεγονός ότι έχουν κάποιες εκατοντάδες επιστραφή, αλλά υπάρχουν δεκάδες αν όχι εκατό, εκατοντάδες χιλιάδες Αφγανοί στις γειτονικές χώρες. η, η κύριε Νάρτ, ε, δεν, όταν μιλάμε για την κυβέρνηση δεν αναφερόμαστε μονάχα στην ε, Καμπούλ. Ε, υπάρχει ε, μία εκπρόσωπος βεβαίως χώρας που ασχολείται πολύ με το Αφγανιστάν που λέει ε, πάντα ότι ασχολούμαστε μόνο με την κυβέρνηση της Καμπούλ. Ωστόσο, εδώ εμείς αναφερόμαστε στο σύνολο του πληθυσμού, κυρίως αυτούς που ζουν στην πρωτεύουσα αλλά και στις ε, πρωτεύουσες ε, των ε, επαρχιών και είναι αλήθεια ότι ο μεγαλύτερος πληθυσμός βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές ενώ εδαφικά μπορεί οι Ταλιμπάν να κατέχουν μεγαλύτερο, μεγαλύτερη επιφάνεια. Υπάρχουν όντως και κάποιες επαφές που άρχισαν περίπου ένα χρόνο πριν με τους Ταλιμπάν είναι γεγονός ότι και οι Ταλιμπάν θα πρέπει να συμβάλλουν με το δικό τους ε, τρόπο ε, και στην ειρήνευση της ε, χώρας και ερχόμαστε σε επαφή με την ηγεσία, όχι απαραίτητα με όλους τους τοπικούς οπλαρχηγούς. Είναι γεγονός ότι το παρελθόν είναι βαρύ, τα λάθη είναι πολλά, ωστόσο είναι γεγονός ε, ότι υπάρχουν αυτοί οι οποίοι βλέπουν την κοινωνία διαφορετικά από ό,τι τη βλέπουμε εμείς, αλλά ε, και αυτοί οι οποίοι έχουν ε, θεμητές προσδοκίες να ζήσουν σε ηρεμία και δημοκρατία. Υπάρχουν θέματα ασφάλειας, θέματα οικονομικά που μας ενδιαφέρουν και μας και δεν είναι δυνατόν να να λέμε ότι οι αφγανικές δυνάμεις θα δουλέψουν για το, υπό τον έλεγχο της Ρωσίας, του Πακιστάν, της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο, μια φόρμουλα ε, που θα επιτρέπει την ειρηνική συνύπαρξη όλων των πληθυσμών. Αυτό είναι γνωστό και από άλλες περιπτώσεις και από άλλες χώρες και λέγεται συμπεριληπτική ε, ειρηνευτική διαδικασία, inclusive peace process. Ε, κύριε ε, Γκάλερ, δεν πρέπει να υποτιμούμε τις ειρηνευτικές διαδικασίες. Αυτές μπορούν να ξεκινήσουν όταν θα υπάρξει κάποια συμφωνία μεταξύ ΙΠΑ και Ταλιμπάν. Αλλά συνολική ε, επίλυση σημαίνει ότι όλες οι πλευρές συνεργάζονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ανέλαβε από τον Απρίλιο του 19, θέλει να παραμείνει δεσμευμένη στο Αφγανιστάν. και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε και τον ρόλο του εγγυητή της ε, διαδικασίας ε, ειρήνευσης. Αυτό άλλωστε είναι κάτι το οποίο έχουμε μεταφέρει και στην πλευρά των ε, Ταλιμπάν. Ίσως να είναι λίγο ιδεαλιστική έτσι ε, θέση. Από την άλλη πλευρά όμως ε, δεν θέλουμε να ξαναμπούμε ε, σε αυτό το χάος το οποίο οδήγησε σε τόσους νεκρούς. Δεν θέλουμε παραπάνω νεκρούς, παραπάνω εκτοπισμένους, περισσότερους μετανάστες πρόσφυγες. Για να γίνει όμως πραγματικότητα αυτό που λέω, χρειάζεται οπωσδήποτε ε, οικονομική βοήθεια. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει να αλλάξουν κάποιες παράμετροι, αλλά δεν είναι δυνατόν να πούμε ας φύγουμε από αυτό το μέρος όσο γίνεται πιο γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ ε, και θα δώσω το λόγο στον κύριο Πιέρ Αμιλχάτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιες παρατηρήσεις που έγιναν σχετικά με την μετανάστευση ή τον εκτοπισμό, ε, αναγκαστικό ή όχι. Το Πακιστάν, το Ιράν, η Τουρκία και το Αφγανιστάν το ίδιο πάντοτε εγνώρισαν στην ιστορία τους τη μετανάστευση. Αυτό που βλέπουμε πρόσφατα, η σημερινή δηλαδή πραγματικότητα, είναι ότι έξι εκατομμύρια Αφγανοί βρίσκονται σήμερα στο Ιράν και στο Πακιστάν. 2,5 εκατομμύρια έχουν απομείνει στη χώρα. Εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια έχουν απομένουν μάλλον στο Πακιστάν μετά τις ε, αναγκαστικές επιστροφές. οι υπόλοιποι που βρίσκονται στο Ιράν έχουν κάποια πρόσβαση σε στοιχειώδεις υπηρεσίες, αλλά χωρίς να τους προσφέρεται η δυνατότητα της υπηκότητας της Ιρανικής. Και πάντοτε υπήρχαν και εποχιακές μεταναστεύσεις μεταξύ Ιράν και Αφγανιστάν, κάτι που βλέπουμε και σε πολλές άλλες χώρες και περιοχές του κόσμου. Το Ιράν δεν διώχνει δεν επιστρέφει μαζικά τους Αφγανούς. 3,5 εκατομμύρια περίπου υπολογίζουμε Αφγανοί ότι βρίσκονται στο Ιράν. Και το 300 δεν είναι τόσο μεγάλος αριθμός, επομένως ίσως είναι στα πλαίσια μιας ε, κανονικής διαχείρισης μετανάστευσης, το να εξηγήσει κανείς αυτές τις επιστροφές δηλαδή. οι σημαντικές επιστροφές από την Τουρκία, το πιο πρόσφατο μέγεθος είναι 200 την ημέρα, που αποστέλλονται με αεροπλάνο πίσω στη χώρα. Εμείς κοιτούμε, παρακολουθούμε τις επιστροφές αυτές προσπαθώντας να βοηθήσουμε συμπεριλαμβανομένων και των Αφγανών που επιστρέφουν από την Ευρώπη. Όλοι οι Αφγανοί που επιστρέφουν από την Ευρώπη είναι ελάχιστοι βέβαια. Και έχοντας χρησιμοποιήσει όλες τις νόμιμες οδούς που διατίθενται στο έδαφος μας. Έχουμε και κάποιους που αρνούνται να επιστρέψουν. Επομένως είμαστε θα έλεγα αυστηροί, αλλά σεβόμαστε και τις ε, διατάξεις του, της νομοθεσίας. Σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχουμε σε αλλοδαπούς να παραμένουν στο εδαφός μας. Για την κοινωνία των πολιτών και την ε, ελπίδα της ανεξαρτητοποίησής της τελικά. Όλα αυτά σχετίζονται και με τη διαφορά μεταξύ των αστικών κέντρων και της Υπέθρου. Στην Υπέθρο προφανώς η παράδοση κυριαρχεί, αλλά σε άλλες περιοχές της χώρας βλέπουμε φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να είναι ιδιαίτερα δραστηριε και βλέπουμε και πολύ θαραλέε προσπάθειες από τις γυναίκε του Αφγανιστάν να πιέζουν για ισότητα, για πρόσβαση στην παιδεία, στην υγεία και για την δραστηριοποίησή τους στον οικονομικό, στο οικονομικό πεδίο και στο πολιτικό πεδίο όπως και στο αθλητικό πεδίο που είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα για αυτές. Έχει σημειωθεί εκπληκτική πρόοδος θα έλεγα, αλλά προφανώς ο δρόμος είναι πάρα πάρα πολύ μακρύς. Εμείς υποστηρίζουμε τις οργανώσεις αυτές με όποιο τρόπο μπορούμε, λέει ο μιλητής. Αυτά θα είχα να πω και νομίζω για την συμπερίληψη της κυβέρνησης του Αφγανιστάν ο Γκούρνερ απάντησε ε, δηλαδή στην ειρηνευτική διαπραγμάτευση αυτό είναι απολύτως απαραίτητο διότι επισήμω είναι η διαπραγμάτευση μεταξύ της κυβέρνησης και άλλων ομάδων γνωρίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Αμερικανών και των Ταλιμπάν ήταν και σχετικά με την συμμετοχικότητα της διαδικασίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ε, τη συμμετοχή στη διαδικασία ε, εθνικών αρχηγών, τοπικών αρχηγών κτλ. Πολεμαρχηγών στην ουσία, σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις. Και το κατά πόσον και αυτοί θα έπρεπε να συμμετάσχουν στην ειρηνευτική διαδικασία. Υπό την έννοια της διεθνούς ανάπτυξης και συνεργασίας δεν είναι κάτι που θα επιθυμούσαμε να δούμε γρήγορα. Γιατί έχουμε δει ξανά και ξανά ότι απλά απαιτούν το δικό τους μερίδιο, τη δική τους πίτα και αυξάνεται διαρκώς η διαφθορά. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους Ευχαριστούμε τον κύριο Βίγκαν και τον κύριο Αμελάτ για την ανταλλαγή αυτή απόψεων. Είναι δύσκολο να καταλήξει κανείς επί τόσο περίπλοκου ζητήματος σε κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για να έχουμε συνεργασία και πρέπει επίση να διοργανώσουμε και άλλε συναντήσεις από αυτού. Πρέπει να συνεχίσουμε να συζητούμε, να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε, να είμαστε βέβαιοι για το ορθό τη πολιτικής μας και για τους πόρους. Σας ευχαριστώ και με αυτό που μπορούμε να κλείσουμε το σημείο. Ο κύριο Μακάλιστερ, ευχαριστώ Τόμας. Προτείνω. Thank you. Thank you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 αν θα μπορούσα να ζητήσω ευγενικά από τους ε, φίλους του αφγανικού θέματος να συνεχίσουν εκτός θεθούσης. Ο κύριος Σικόρσκι Γκοσμποντίν ή λάθος το είπα. Πάνιε, μάλιστα. Λοιπόν, μαζί με τους φίλους και συναδέλφους της Επιτροπής ΔΕΒΕ έχουμε το σημείο 11 για τη θέσπιση μηχανισμού γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας, NDICI, το αγαπημένο μας θέμα, και μέσον. Είχαμε ένα πρώτο γύρο διοργανικών συζητήσεων 23 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. Επ' αυτού θα έχουμε ενημέρωση και θα ζητούσα τους συνεισηγητές να μας δώσουν μια σύντομη επισκόπηση του, των θεμάτων που συζητήθηκαν στον πρώτο αυτό τριμερή διάλογο με Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πω ότι είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις γιατί όλοι συμμερίζονται το στόχο της επίτευξης ε, συμφωνίας το συντομότερο δυνατόν ώστε να τεθεί σε ισχύ αυτή, αυτός ο μηχανισμός το συντομότερο δυνατόν κατέστη βέβαια σαφές ότι δεν είμαστε έτοιμοι να υποχωρήσουμε επί της ουσίας λόγω της χρονικής πίεσης. Προτού δώσω τον λόγο στους συνεισήγητες. θα δώσω τον λόγο στον κύριο Τομπέ, ως πρόεδρο της ε, ΔΕΒΕ, και έχουμε και NDCI και ΙΠΑ που συνδέονται στενά και θα δώσω και στους συνεισηγητές επί του μέσου αυτού το λόγο, αλλά ας ακούσουμε NDICI πρώτα και μετά EPA. Αν συμφωνητές πάνω μισή ώρα έχουμε, Τόμας. Ευχαριστώ, David. Να τονίσω και εγώ από την πλευρά μου τη σημασία που έχει το θέμα αυτό για τις επιτροπές μας και το γεγονός ότι ως Κοινοβούλιο στείλαμε το μήνυμα στα άλλα δύο θεσμικά όργανα ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις, κάτι που είναι αναγκαίο δεδομένη της περιπλοκότητα του θέματος και τη ε, άμεση έναρξης ε, εφαρμογής του νέου ΠΔΠ. Έχουμε πει πολλέ φορέ ότι πρέπει να οριστικοποιήσει το Συμβούλιο τη θέση του για το ΠΔΠ προτού μπορέσει το Κοινοβούλιο να εξετάσει το περιεχόμενό του και να ε, καθορίσει τη στάση του εν ώψη των διαπραγματεύσεων. Χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή θα έλεγα να δώσουμε το λόγο στους συνεισηγητές για να μας ενημερώσουν σχετικά με τον τριμερή διάλογο. Έτσι θα το κάνουμε λέει ε, ο κύριος Μεκάλιστερ, ο κύριος Γκέρενς έχει φύγει οπότε το λόγο θα πάρει ο κύριος Γκάλερ. Συνάδελφοι, Χαιρόμαστε και εμείς πολύ για την, ε, για την δυνατότητα που είχαμε να ξεκινήσουμε επιτέλους τις διαπραγματεύσεις ε, με τον, ε, ως συνομοθέτης, με παράγοντα διευκόλυνση στην Κομισιόν που θα, καθορίσει πλέον, θα καθορίσουν πλέον την διαμόρφωση αυτού του ταμείου, αυτού του μηχανισμού με προϋπολισμό 90 δισεκατομμύρια για, τα, για την 7 ετία του πι δελτα πι. Ε, ξεκινήσαμε λοιπόν τις διαπραγματεύσεις, ήμασταν εμείς οι συνεισηγητές, οι πρόεδροι των επιτροπών, ε, καθώς και οι εκπρόσωποι των ε, επιτροπών ΦΑΜ και ΜΠΑΤΖ, μαζί με τους σκιώδεις και τους συντονιστές των επιτροπών μας. Είχαμε επίσης μαζί μας τον πρέσβη της Φιλανδίας εκ μέρους του Συμβουλίου. Επικεφαλής της Αντιπροσωπής Κομισιόν ήταν ο κύριος ε, Νίμιτσα, Επίτροπος Αρμόδιος για θέματα διεθνούς συνεργασίας. Έγιναν κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις, ε, περιγράφηκαν οι προτεραιότητες και οι επιδιώξεις μας. Ακόμη δεν έχουμε μπει στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά το κείμενο του κανονισμού αυτού καθεαυτού. Όμως με χαρά μπορούμε να σας ανακοινώσουμε ότι έχουμε συμφωνία επί των ε, μεθόδων εργασίας και ε, έχουμε και ένα χρονοδιάγραμμα έως το τέλος του χρόνου. Θα προχωρήσουμε κατά ομάδες θεμάτων και θα αξιοποιήσουμε ε, την καλή δυναμική που υπάρχει σε πολλά θέματα και στη συνέχεια θα πάρουμε τα πιο ακανθόδη θέματα. Θα, στόχος είναι να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία θα τεθεί στη ψηφοφορία και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Είχαμε εντολή, ε, δώσαμε μάλλον εντολή και στο τεχνικό προσωπικό ώστε να ε, καταρτήσει ένα τεχνικό κείμενο το οποίο θα συζητηθεί στις 5 Δεκεμβρίου με το οποίο ελπίζουμε να συμφωνήσουμε επί των ουσιδών θεμάτων του κανονισμού. Στο πλαίσιο αυτό τα μέλη της Επιτροπής θα λάβουν τα προσωρινά ε, συμφωνηθέντα με ε, τη μορφή ενός τετράστιλου εγγράφου και θα γίνουν και ε, αντίστοιχες ενημερώσεις όπως η σημερινή μετά από κάθε γύρο διαπραγματεύσεων. Επίσης υπάρχει κοινή αντίληψη ότι ε, το, ο τίτλος του κανονισμού είναι με περιττό τρόπο περίπλοκο και θα πρέπει να δοθεί ένας πιο απλός τίτλος. Αυτό όμως μάλλον θα γίνει στο τέλος των διαπραγματεύσεων αφού θα έχει καθοριστεί το περιεχόμενο του κειμένου. Πάντως κάθε πρόταση προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ευπρόσδεκτη. Καθώς υπάρχουν μια σειρά από οριζόντιες διατάξεις στην εντολή μας για το NDICI που είναι ε, ε κοινέ με τη θέση του Κοινοβουλίου για, την, ε, για τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας, το IPA 3, όπως είπατε κι εσείς, Έχουμε ε, ε, εκπροσώπους του Κοινοβουλίου από τους Σοσιαλιστές και, τους, ε, και το ΕΛΚ που θα συμμετάσχουν σε όλη τη διαδικασία ε, της διαπραγμάτευσης. Αυτά από τον κύριο Γκιόρενς. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ, λέει ο πρόεδρος. Ποιος άλλος θα ήθελε το λόγο. Οι συνεισαγητές, η κυρία Μαρία Αρένα. Ευχαριστώ Μάικλ για την παρουσίαση της διαδικασίας σε σχέση με την διαπραγμάτευση και τον τριμερή διάλογο. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι ε, στο Κοινοβούλιο βεβαίως κατανοούμε ε, την ε, σημασία του θέματος, αλλά κατανοούμε και την δυσκολία της συζήτησης που έχουμε απέναντί μας από τη στιγμή που διήστανται οι απόψεις του Συμβουλίου της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπενθυμίσαμε βεβαίως τις αρχές που είναι σημαντικές ε, στην θέση του Κοινοβουλίου. Πρώτον, ε, ε, σωστή και ουσιαστική εμπλοκή του Κοινοβουλίου στις στρατηγικές επιλογές και όσον αφορά την ε, ε, συνήθη διαδικασία και όσον αφορά και τις έκτακτες αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνονται ε, σε επίγουσες καταστάσεις. Δεύτερον, ο λόγος που πρέπει να έχει το Κοινοβούλιο στην μελλοντική ε, ε, στον μελλοντικό προγραμματισμό και τρίτον απλούστευση των εργαλείων παρέμβασης. Άρα δεν χρειάζεται να κατακαιρματιστεί ε, η πρόταση που έχει διατυπωθεί μέχρι τώρα. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν όπως ανέφερα αποκλίνουσα απόψεις αλλά υπάρχουν και στοιχεία σύγκλησης ανάμεσα στις θέσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έστω και αν πρόκειται για μερική κο ε, μερική εντολή από πλευρά του Συμβουλίου, κυρίως όσον αφορά τα προγράμματα εκρίζωση της φτώχεια. Ε, κατά την έννοια αυτή, το Κοινοβούλιο θα ε, εγκρίνει και θα υποστηρίξει τους διάφορους δείκτε. Ε, επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της δημοσιας αναπτυξιακη αναπτυξιακής βοήθειας από 92-95%, καθώς επίσης και το ποσοστό του ΑΕΠ στην αναπτυξιακή βοήθεια. Επίσης, προτείνω προτείνουμε ε, να ε, ε, χρηματοδοτηθεί με 45% του εργαλείου το θέμα της για το περιβάλλον ε, και 85% για τις δράσεις ε, όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε την καλή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, τα ε, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμείς θέλουμε μια συγκεκριμένη ρήτρα η οποία θα συμπεριλάβει και την πυρηνική ασφάλεια. Νομίζω ότι είναι σημαντικό εδώ ε, να αναφερθεί η θέση του Κοινοβουλίου στην πρωτοβουλία που ανέλαβε την προηγούμενη εβδομάδα στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο Ράζα Γιουνεβιτσιάν έχει θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ και τους δύο Προέδρους. Θα πω κάποια λόγια για ορισμένα από τα θέματα που έχουμε συζητήσει ήδη. Όσον αφορά τη δομή, τη διάρθρωση του πεδίου εφαρμογή και τον προπολογισμό. Σε πρώτη ανάγνωση, ανάγνωση, το Κοινοβούλιο συμφώνησε με την πρόταση ενσωμάτωσης όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων υπό τον ε, γεωγραφικό πυλώνα ε, με ομαδοποίηση θεματική ε, και με αντίστοιχη αποθεματοποίηση. Όσον αφορά τα χρήματα, εμείς υποστηρίξαμε την αύξηση ε, στα 93 δισεκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδοτική βοήθεια προς την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, καθώς και την πρόβλεψη συγκεκριμένων ε, κονδυλίων για την Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική. Για την Αφρικανική ε, Ήπειρο, ε, καθώς και για το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που θα κάλυπτε Αφρική και Καραϊβική. Ε, επίσης, προτείναμε την αύξηση του θεματικού πυλώνα με ε, ενίσχυση των κονδυλίων για τις οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσον αφορά το παγκόσμιο πρόγραμμα που αφορά κυρίως τη βιώσιμη ανάπτυξη, εμείς καλέσαμε να υπάρξει ε, χρηματοδοτική ενίσχυση του προγράμματος αυτού ε, με αύξηση από 3 δισεκατομμύρια σε 4,5 δισεκατομμύρια. Για το EFSD ε, το Κοινοβούλιο υποστήριξε την ένταξη του νέου EFSD Plus στο NDICI και τη δημιουργία ε, ε, ε μιας ε, ενιαίας εγγύης εξωτερικής δράσης. Υποστηρίξαμε επίσης τη συνέχιση των δράσεων της ΕΤΕΠ στο εξωτερικό με ε, ενίσχυση της εξωτερικής τάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ το Κοινοβούλιο πρότεινε να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό ε, παράθυρο επενδύσεων με δυνατότητα τουλάχιστον ενός δισεκατομμύριου ευρώ που θα εφαρμόσει η ΕΤΕΠ. Το Κοινοβούλιο επίσης από το τρέχον EFSD χρησιμοποιεί ε, τα αποθεματικά που έχει το Ταμείο αυτό προκειμένου να ενισχυθούν ανθρώπινα δικαιώματα και νομίζω ότι και η Επιτροπή μας έκανε μια ε, ad hoc επίσκεψη στην Αιθιοπία και η διεισόμαση διαπίστωσε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Επίσης το Κοινοβούλιο υποστήριξε την διεύρυνση της ε, γεωγραφικής κάλυψης του FSD EFSD+, ε, σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και της γειτονίας για κατά προτεραιότητα ε, προώθηση εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, και ίσως το πιο σημαντικό, που ανέφεραν και, ανέφερε και ο κύριος Γκάλερ, ορισμένοι πιστεύουν ότι το να βαφτίσεις ένα μωρό είναι πολύ σημαντικό για το, το τι όνομα θα δώσεις, είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή που θα ζήσει ο άνθρωπος αυτός. Αν το όνομα του δεν είναι κατάλληλο, τότε θα αποτύχει στη ζωή του. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να διαλέξουμε με προσοχή το όνομα γι' αυτό το μωρό μας και πιστεύω ότι ε, θα πρέπει ο τίτλος να αντικατοπτρίζει την απλότητα ε, και την αποτελεσματικότητα που θέλουμε να προσδώσουμε σε αυτό το μηχανισμό που όνομα το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να είναι το NDICI. Σας ευχαριστώ. Σχόλιο. Και καλό όνομα να βρούμε για το μωρό. Φαίνεται ότι έχουμε την ε, ανόητη ικανότητα να καταστρέφουμε τα πάντα μέσω τελείως ανόητων ακρονίμων. Θα δώσω τώρα το λόγο στον ε, Μίχαλ Γκάλα, γιατί καταρχάς τοποθετήθηκε εξ ονόματος του κύριου Γκέρν. Σε ευχαριστώ πρόεδρε, σύντομα και επί της εμείς παρουσιάσαμε την πρώτη ε, τοποθέτηση του Κοινοβουλίου, Πρώτη ανάγνωση δηλαδή, το Συμβούλιο τον Ιούνιο και ακολούθως το Σεπτέμβριο, κάποια στοιχεία κατά την άποψή μας ουσιαστικότατα, εξαρτώνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, ως τμήμα των διαπραγματεύσεων του ΠΔΠ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το Μάρτιο του χρόνου Κάτι που φοβούμε θα είναι υπό τη Γερμανική Προεδρία, λέει ο κ. Γκάλα. Και στι 10 Οκτωβρίου ζητήσαμε από την Επιτροπή σχέδιο ε, εκτάκτου ανάγκης για την ε, τυχόν παράταση του υφιστάμενου μηχανισμού για να μην έχουμε πλέον τη χρονική πίεση που θα μας απέτρεπε να επιτύχουμε το στόχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίση υποστηρίζουμε την, Επιτροπή, την πρόταση Επιτροπή για τη συγχώνευση των δημοσιονομικών μέσων και του μηχανισμού γειτονία, που είναι υπό συγκεκριμένο κεφάλαιο του κανονισμού, Όπω και για το Ταμείο Ευρωπαϊκή ανάπτυξη, που ήταν πάγιο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό θα δημιουργούσε μια μόχλευση πολιτική πολύ πιο αποτελεσματική και επιφανή, εμφανή, όπως και προσθέμενη αξία έναντι τη παρούσα κατάστασης και θα ομοδοποιούσε κάποιες παράλληλες ε, διαδικασίες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και βεβαίω ε, θα πρέπει να στηρίζει το μέσο τον μελλοντικό, το μελλοντικό πλαίσιο πολιτική και όχι αντίστροφα. Πάντως επί των ουσιαστικών αυτών δύο μέσων, γειτονίας και αναπτυξιακού, εμείς θεωρούμε ότι αυτά είναι μέρος της παρούσας νομοθετικής διαδικασίας και επομένως θα υπόκειται σε μελλοντικέ διαπραγματεύσεις τριμερού διαλόγου. Δηλαδή είχαμε προειδοποιήσει να μην θεωρηθεί ότι πρόκειται για τετελεσμένο και το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μπλοκάρισμα της διαδικασίας. και εγώ είμαι υπέρ ε, του κοινού παρανομαστή ε, της απλής πρότασης για το όνομα του ε, μέσου να είναι το Global Instrument το οποίο λέει ο κύριος Μακάλιστερ σύντομα θα είναι το GI προφανώς Μάρκ Ταραμπέλα παρακαλώ Ευχαριστώ πρόεδρε Σύντομα ήθελα να τοποθετηθώ αλλά σε γενικούς όρους έχοντας ακούσει τον κύριο Γκάλα και τους του κύριου Γκέρνς και την κυρία Ρίνα, νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να είμαστε ελέγγυοι σε αυτό το κοινοβούλιο, διότι είχαμε φιλόδοξη στάση πέρσι το, το Μάρτιο, να θυμίσουμε. Και ε, όπως πολύ συνήθως συμβαίνει, ανεξαρτήτως αρμοδιοτήτων, είτε η Επιτροπή είτε το Κοινοβούλιο είναι η πιο φιλόδοξη και τελικά η Κομισιόν έρχεται να φρενάρει άπαντες. και το οποίο μπορεί να είναι καλό τρίκ στη Νέα Υόρκη στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά όταν μιλούμε για πραγματικά προβλήματα είμαστε πολύ λιγότερο αποτελεσματικοί. Πρέπει να υποστηρίξουμε τον συνεισηγητή και να διατηρήσουμε τη φιλόδοξη θέση μας. Γιατί πολλοί άριθμοι φορείς που ασχολούνται την καταπολέμηση της ένδυας, ε, την κλιματική αλλαγή κτλ. και διάφορες προσπάθειες αναπτυξιακές, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη στιγμή αυτή και να είμαστε αλληλέγγυοι και φιλόδοξοι. Τώρα, η πρώτη συναντήση η δεν δίνει τίποτα. Οι τεχνικέ που έχουμε σήμερα δεν μας διασφαλίζουν καθόλου για την θέση του Συμβουλίου. Από αυτά που έχω διαβάσει για τη χθεσινή συνάντηση δεν πήγαν πολύ καλά τα πράγματα και πάλι το Συμβουλίο έρχεται να ασκήσει, το, να διαρματίσει το ρόλο τροχοπέδης που επιθυμεί, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να διατηρήσουμε τη θέση μας φιλόδοξη. Ευχαριστούμε κύριε Ταραμπέλα. Όταν ζουν, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα επανέλθω στα λόγια του συναδέλφου Ταραμπέλα. Να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές για το θετικό τους πνεύμα. Σε πολλά επίπεδα έχουμε μια φιλόδοξη πρόταση από πλευράς Κοινοβουλίου και πιστεύω ότι μάλιστα ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην καταπολέμηση κλιματική αλλαγή και τα θέματα ισότητας των φύλων. Κάναμε πολύ καλή δουλειά για να διαμορφώσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου και τώρα από εμά εξαρτάται να διαδραματίσουμε το ρόλο που πρέπει. Γιατί όπως έλεγε και ο Μάρκ, η φιλοδοξία του Κοινοβουλίου είναι πάντοτε η και μετά κατέρχεται, αλλά αυτό το μέσον πραγματικά πρέπει να δώσει αποτελέσματα στην κλιματική αλλαγή και στην ισότητα των φύλων στις εξωτερικές μας παρεμβάσεις. Έχουμε ρόλο εδώ να διαδραματίσουμε και ήθελα να επιμείνω επίση κάτι που ανέφερε και η κυρία Ρενά, το θέμα της διακυβέρνηση. Νομίζω ότι στο παρελθόν αυτό το μέσον είχε απόλυτη έλλειψη κενό κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αυτό το βελτιώσαμε σε ουσιαστικό βαθμό αλλά είναι ένα από τα ζητήματα που θα είναι τα πιο αντιφατικά με την Επιτροπή και με το Συμβούλιο. Και εδώ πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εγγυηθούμε και την ευελιξία για την εκτέλεση του μέσου, αλλά και έναν κοινοβουλευτικό έλεγχο. Γιατί είναι και τα δύο αυτά σημαντικά. Υπό την έννοια αυτή, ή μάλλον και σε αυτό το επίπεδο είμαστε φιλόδοξοι, πρέπει όμως να υπερασπιστούμε τη θέση μας, γιατί είναι ένα από τα σημεία στα οποία το νέο μέσο μπορεί να έχει ουσιαστικότατη βελτίωση. Κοινοβουλευτικού δηλαδή ελέγχου. Ευχαριστώ και πάλι τους συνεισηγητές. Ευχαριστούμε. Συνάδελφοι, υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο? Όχι από ό,τι βλέπω. Οπότε, όπως έχω ήδη ανακοινώσει, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους δύο συνεισηγητές μας για το ΙΠΑ. που, είναι, που μοιράζεται το ίδιο, την ίδια αγγλική συντομογραφία με το διεθνές φωνητικό αλφάβητο. Αλλά για εμά, εμείς εδώ θα μιλήσουμε για το μηχανισμό προνταξιακής βοήθειας. Να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Ζόφκα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την περιφερειακή σταθεροποίηση. Εμείς αποφασίσαμε να αναβάλουμε τις διαπραγματεύσεις ελπίζοντας να αναλάβει τα καθήκοντα της η νέα Κομισιόν, ο νέος επίτροπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κατάλληλη συμφωνία. Η διαπραγματευτική ομάδα λοιπόν πήρε την ε, απόφαση να αναβάλει ε, την ε, πρώτη διαπραγμάτευση που είχε προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου. Ο αποκλεισμός σημαντικών στοιχείων από το νομοθετικό κείμενο ε, από το Συμβούλιο θεωρούμε ότι είναι τελείως απαράδεκτος. Και αυτό ισχύει ιδίω για τις διατάξεις που θεωρούμε ότι αφορούν το ΙΠΑ, όπως είναι οι απαιτήσει για την επικοινωνία και την ορατότητα. Δεύτερον, η διαπραγματευτική ομάδα θέλει να καταλήξει σε διοργανική συμφωνία σχετικά με τις λεπτομέρειες για την επικαιροποίηση των παραρτημάτων του ΙΠΑ οι συνομοθέτες δεν μπορούν να γνωρίζουν πόσο λεπτομερή θα πρέπει να είναι τα παραρτήματα αν δεν υπάρχει συμφωνία για το αν θα επικυροποιούνται μέσω κατεξουδότηση πράξης ή μέσω ε, ολοκληρωμένης νομοθετικής διαδικασίας. Αυτά από μένα. Να δώσω το λόγο στο συνεισηγητή μου, τον κύριο τον Πίτσουλα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, να προσθέσω και εγώ δύο παρατηρήσεις στα όσα μας ε, είπε ήδη η κυρία Ζόφκο. Θεωρούμε και εμείς ότι οι διαπραγματεύσεις για, την, για το επικαιροποιημένο πλαίσιο για την πρωταξιακή χρηματοδότηση 2021 έως 2027 θα πρέπει να διεξαχθεί μετά την ανάληψη των καθηκόντων της ε, νέας Επιτροπής. Και παρά το γεγονό ότι η Κομισιόν είναι απλώ ένα διευκολυντή, εμεί είμαστε πεπισμένοι ότι το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση τη ε, διεύρυνση θα πρέπει να συζητηθεί με τον νέο Επίτροπο. Και τέλο θέλω να ολοκληρώσω λέγοντα ότι αυτή τη στιγμή αναζητούμε πιθανή ημερομηνία για την πρώτη συνάντηση τριμερού διαλόγου που θα μπορούσε να βρίσκεται κάπου στα μέσα του Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρο. Συνάδελφοι, υπάρχει κάποιο που θα ήθελε το λόγο. Υπάρχουν ερωτήσει, παρατηρήσει, σχόλια από πλευρά σα όσον αφορά το είπα. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Και έτσι νομίζω ότι ολοκληρώσαμε την σημερινή μας συνεδρίαση. Να σας ευχαριστήσω. Συγγνώμη, τι. Α, ναι. Να ευχαριστήσω καταρχάς τους συναδέλφους από την Επιτροπή ΝΤΕΒΕ, ιδίως τον Τόμας και τώρα προχωράμε στην συνεδρία συντονιστών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Μόνο οι έχοντες εργασία παρακαλώ να μείνουν εδώ, όλοι οι άλλοι να αποχωρήσουν. Καλό σας βράδυ.